μια ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τότε πραγματικά όλοι θα κερδίσουν από τέτοια συμφωνία. Ευχαριστώ πολύ, Επιτρόπε. Ευχαριστώ όλου που συμμετείχαν στην συνεδρίαση. Η ψηφοφορία θα εξελιχθεί στην επόμενη περίοδο συνόδου. Το επόμενο θέμα στη σημερινή συνέντευξη είναι η προβολική ερώτηση προ την Εκκλησική Επιτροπή όσον αφορά τη στρατηγική για την περιοχή του Ατλαντικού. Ο κ. Κάντεκ έχει το λόγο. You want... Can I Mr. Kadek, sorry. Alain, deux secondes. Μισό λεπτό, Alain. Do you want the floor? Παρακαλώ, θέλετε το λόγο, κυρία μου. Nothing, nothing else. I'm sorry. Okay, fine. Please, Alain. Όχι, ευχαριστώ. Ωραία. Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχήν ευχαριστώ την Επίτροπο Δαμανάκη που είναι παρούσα σήμερα για να απαντήσει στην προφορική αυτοερώτηση για τη στρατηγική για την περιοχή του Ατλαντικού. Το 2010 το Συμβούλιο ζήτησε από την Εκκλησία Επιτροπή να προετοιμάσει μια ευρωπαϊκή πολιτική για την περιοχή του Ατλαντικού μέχρι το 2011. Με, ζει με άλλου συναδέλφου, ε, ανέλαβα την πρωτοβουλία να προετοιμάσω μια προφορική ερώτηση προ την Εκκλησική Επιτροπή μια προφορική ερώτηση που υπεγράφηκε από πάνω από 50 βουλευτές από όλες τις ε, πολιτικές ομάδες και θέλω να σας ευχαριστήσω για την υποστήριξη. Ταυτόχρονα θα υποβάλλεται αυτή η ερώτηση εξ ονόματο της Επιτροπής Περιφερικής Ανάπτυξης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τις πολιτικές ομάδες για την εργασία τους που επέδεψαν ευρεία συνένεση. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που συνέβαλαν στον εμπλουτισμό του κειμένου αυτού με τις τροπολογίε του. Η περιοχή του Ατλαντικού χαρακτηρίζεται από ιδιάζοντα χαρακτηριστικά. Πρόκειται για ένα πολύ δυναμικό χώρο, θαλάσσιο χώρο. Ταυτόχρονα είναι μια λεπτή περιοχή όσον αφορά το περιβάλλον που θα πρέπει να διατηρήσουμε. Ένα περιβάλλον που πλήττεται από τις κλιματικές αλλαγές. Είναι μια περιφερειακή περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χαρακτηρίζεται από προβλήματα προσβασιμότητας και <clears throat> από το κινδύνο από μεγάλα κέντρα. Γι' αυτό η προβληματική ξεπερνάει τα, τα εθνικά σύνορα και θα πρέπει να βρεθεί η λύση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το ψήφισμα λοιπόν ζητά η στρατηγική για τον αθλητικό να είναι ε, ολοκληρωμένη, το υπόψη και τι και τις ε, εδαφικές ε, πτυχές. Οι περισσότερε είναι στρεμμένες προ τη θάλασσα. Θα πρέπει λοιπόν να ενθαρρυνθούν οι κοινέ σχετικέ πολιτικέ. Η εδαφική διάσταση αφορά την ανάπτυξη αστικών κέντρων, περιφερειακών κέντρων και γενικά η στρατηγική για την περιοχή του Ατλαντικού θα πρέπει να ενταχθεί σε μια εδαφική πολιτική, πολιτική σύνοχης ολοκληρωμένης και περιφερειακής προσέγγισης. Θα πρέπει καλύτερα να συντονιστούν οι διάφορες πολιτικές και όσον αφορά συγκεκριμένες προβληματικές. Η στρατηγική αυτή θα πρέπει να ανοιχτεί σε όλες τις περιοχές της, Γαλλικής, Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν όρια στον Ατλαντικό. σε της Μακρονησίας. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τις εξωτερικές πτυχές στρατηγική όσον αφορά το θέμα της ασφάλειας και τα θέματα των διεθνών εμπορικών σχέσεων. Η στρατηγική για τον Ατλαντικό θα πρέπει να βελτιώνει την προσέγγιση και να προσανατολιστεί στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2020, μετά το 2014 δηλαδή. Δεν θέλουμε να δαπανίσουμε περισσότερα, αλλά να δαπανίσουμε καλύτερα, εστιώνοντας τις ε, λόγω πολιτικές στον Ατλαντικό. Θα πρέπει λοιπόν η στρατηγική να προσανατολίζεται πολύ καλύτερα στην περιφερειακή πολιτική και στα λάσια πολιτική, να αναζητήσουμε συνέργειες με άλλες πολιτικές όπως παραδείγματος χάνει τα ευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, την κοινή πολιτική αλληλεία, τουρισμό, πολιτική περιβάλλοντος, πολιτική ενέργειας ή και το πρόγραμμα πλαίσιος έρευνας και ανάπτυξης. Η στρατηγική αυτή θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ από το 2014 και να συνοδεύεται από πολιετές ε, χρηματοπιστωτικό πλαίσιο. Θα πρέπει ιδίω να υπάρχουν ε, πολιτικές για να μην υπάρχει αποκλεισμός. Θα πρέπει να αναπτυχθεί η θαλάσσια πολιτική που θα ευνοήσει ιδιαίτερα τι αναλόγες Θα πρέπει ταυτόχρονα να ενδυναμωθεί η διάσταση βορρά-νότου στον Λατικό, εφαρμόζοντας αυτοκινητό δρόμους της θάλασσας από την Ανταλουσία μέχρι τη Σκοτία. Θα πρέπει ταυτόχρονα να δούμε τι γίνεται με τι μεταφορέ από Ανατολή προς Δύση, ιδίως στις δρομικές μεταφορές μεγάλη ταχύτητα. Θα πρέπει να υπάρχει μια συγκεκριμένη πολιτική για το συντονισμό με τις πολιτικές ε, της Ευρώπης μετά το 2013. Θα πρέπει να εμπλαχθούν οι ενδιαφορεόμενοι, ιδίως η τοπική και περιφερειακή ε, αυτοδιοίκηση και οι οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών. Η συνεργασία στον τομέα τη για το ελληνικό θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις επιτόπου ανάγκες. Οι προτεραιότητες πολιτικής που θα οριστούν θα πρέπει να είναι αντικείμενο συνένεσης. Η ομάδα της Ευρώπη για την ε, ε, περιφερειακή συνεργασία θα πρέπει να έχει μια ιδιαίτερη διάσταση για τον Ατλαντικό. Αυτά με δύο λόγια οι σκέψει για αυτή τη στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα είμαστε προσεκτικοί όσον αφορά τι εξελίξει τη Εκτελεστική Επιτροπή και θα υποβάλουμε συγκεκριμένε προτάσει. Κύριε Επίτροπε, μπορείτε να διευκρινίσετε ποιε είναι οι προτεραιότητε τη Εκτελεστική Επιτροπή και πώ προβλέπετε να εφαρμοστεί η στρατηγική αυτή και κατά πόσο μπορείτε να λάβετε υπόψη τι ε, απόψει της, ε, του Κοινοβουλίου. Βέβαια, κύριε Πρόεδρε, στο Στρασβούργο βρισκόμαστε. Επαναλαμβάνω. Η κυρία Δαμανάκη. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Καντέκ για αυτή την πρωτοβουλία. Επίσης είναι ευπρόσδεκτες οι ιδέες του. Ευχαριστώ και τα μέλη του Κοινοβουλίου που προσυπέγραψαν την προφορική αυτή ερώτηση. Πλέον εργαζόμαστε για την προετοιμασία μιας θαλάσσιας στρατηγικής για την περιοχή του Ατλαντικού. Πρέπει να σας ε, ενημερώσω ότι είμαι αποφασισμένη να εφαρμόσω μια καλά στοχευμένη στρατηγική ώστε οι θαλάσσιες υποθέσεις να μπουν στην κορυφή των θεμάτων της περιοχής. Βεβαίως παραδέχομαι ότι αυτή η περιοχή έχει μια μεγάλη κληρονομιά σημαντικής περιβαλλοντικής σημασίας και όπου υπάρχουν πολλοί εμπλεκόμενοι έχω ενθαρρύνει όλους αυτούς τους εμπλεκομένους συμπεριλαμβάνουν τις ε, παράκτιες και θαλάσσιες περιοχές του Ατλαντικού ε, να στηρίξουν ενεργά τη στρατηγική αυτή. Ήδη έχουν δείξει μια καλή υποστήριξη στη διάρκεια της προετοιμασίας. Θα συνεχίσω να τους ενθαρρύνω να εμπλέκουν πλήρως την διαδικασία έγκρισης της, πράγμα που θα αποτελέσει κρίσιμο στοιχείο της επιτυχίας της στρατηγικής. Τι μας έχει δείξει μέχρι στιγμής η δημόσια διαβούλευση έδειξε ότι υπάρχει ατλαντική ταυτότητα. Επίσης έδειξε ότι οι εμπλεκόμενοι θεωρούν θετική μια προσέγγιση που να λαμβάνει υπόψη την γεωγραφική, δημογραφική και οικονομική τους ιδιαιτερότητα. Στηρίζουν επίσης τα μέτρα που φέρνουν κοντά τα ε, παράκτια κράτη ε, για θέματα θαλάσσιων ε, γνώσεων την παρακολούθηση της θάλασσας και άλλα. Άρα η αντίδραση που είχαμε στη διάρκεια της διαβούλευσης μας επέτρεψε να θεσπίσουμε προτεραιότητες δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τομέα της ανάπτυξης της περιφέρειας τους ερχόμενους, τους ερχόμενους μήνες. Η στρατηγική του Ατλαντικού θα θεσπίσει συγκεκριμένους στόχους πολιτικής προσφέροντας μια διασταύρωση όλων αυτών των θαλασσίων τομέων. Βασική προτεραιότητα θα αποτελέσει η δημιουργία θέσεων εργασία στην περιοχή. Αυτό απαιτεί πλήρη δέσμευση και ενεργό συμμετοχή των κρατών μελών από τη διάσκεψη των περιφερειακών θαλασσίων περιοχών, των περιοχών της του Ατλαντικού και της θαλά, τους θαλάσσιους οικονομικούς κλάδους. Θα πρέπει οι ευρωβουλευτές να ασχοληθούν με το θέμα αυτό στις περιφέρειές τους. Πράγμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κυρίες και κύριοι, για να εξασφαλίσουμε ότι το θέμα αυτό θα έρθει στο προσκήνιο όσο το δυνατόν περισσότερο, προτείνω η έγκριση να γίνει μετά τη συζήτηση και για την κοινή ελληνική πολιτική. Έτσι θα εξασφαλίσουμε την απαιτούμενη έκθεση σε αυτή την ε, πρωτοβουλία και θα δοθεί και η νέα διάσταση στη νέα αναθεωρημένη αλληλευτική πολιτική πρέπει βεβαίως να ληφθεί πλήρως υπόψη η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και γι' αυτό κύριε Πρόεδρε πιστεύω ότι η Ατλαντική Στρατηγική θα βοηθήσει πρώτον την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της απασχόλησης στην περιοχή μέσω ερευνητικών προγραμμάτων και προγράμματων ε, ε, περιφερειακής ανάπτυξης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον θα επιτευχθούν οι στόχοι της αναθεωρημένης κοινή αλληλεπτική πολιτική και τρίτον θα επιτευχθεί πρόοδος στην προστασία του περιβάλλοντος ενώ ταυτόχρονα θα αναπτυχθεί η θαλάσσια οικονομία με βιώσιμο τρόπο στην ζωτική αυτή σημασία περιοχή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Ρόι για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συγχαρητήρια για αυτή την πρωτοβουλία, η οποία έρχεται την κατάλληλη στιγμή και να ευχαριστήσουμε και την Επίτροπο για τις πρωτοβουλίες της για την θαλάσσια στρατηγική. Εξετάζοντας προσεκτικά το κείμενο, θα πρέπει να σταθούμε σε όλες τις πτυχές τις οποίες θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε από κοινού. Αν κατάλαβα καλά, δεν προσπαθούμε να δημιουργήσουμε νέες δομές. Θέλουμε απλώς οι περιοχές οι οποίες βρίσκονται στις ακτές του Ατλαντικού και αυτές που βρίσκονται στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού θα να έχουν μια ολοκληρωμένη πολιτική για να μπορέσει να υπάρχει ε, μία ε, νέα μέση οδός μεταξύ κρατών μελών και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή είναι η προκαταρκτική μου παρατήρηση. Αν δούμε όμως τις ε, πτυχές και τις ε, διαστάσεις της ε, θαλάσσιας πολιτικής, υπάρχει το θέμα των μεταφορών που έχει περιβαλλοντικές συνέπειες, οικονομικές συνέπειες. Μας ενδιαφέρει και η βιώσιμη ανάπτυξη στα πλαίσια της στρατηγικής 2020, οι ενεργειακές προκλήσεις. Πρόκειται για στοιχεία τα οποία από κοινού επισημαίνουν πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στις ακτές του Ατλαντικού ώστε να μπορέσουν να αναπτυχθούν στο μέγιστο οι δυνατότητές τους. Εγώ προέρχομαι από τις κάτω χώρες, εκπροσωπώ τις κάτω χώρες εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γνωρίζουμε ότι Υπάρχει μια στρατηγική για τη Βαλτική θάλασσα, υπάρχει για τον Ατλαντικό και για τη Μεσόγειο μια ε, στρατηγική, μια στρατηγική για το Δούναβι και τι λείπει. Η Βόρεια θάλασσα. Αν σκεφτούμε τις μακροπεριφέρειες, θεωρώ κυρία Επίτροπε ότι αυτό θα πρέπει να είναι το επόμενο βήμα. Θα πρέπει λοιπόν να έρθει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μία εβδομάδα εδώ στην περιοχή και να μας πείτε τι ακριβώς σκοπεύετε να κάνετε. Μπορείτε να μου δώσετε μια απάντηση. Ο κύριος Κορτές Λάστρα, για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η περιοχή η στρατηγική του Ατλαντικού ενέπνευσε και άλλες περιοχές, τις παράκτητες περιοχές του Δούναβη ας πούμε. Στην περιοχή μου, στην Ισπανία, στο Καντάμπρε από το 1989 συνεργαζόμαστε στα πλαίσια της Σύμβασης των Θαλάσσιων Περιφερειακών Περιοχών με στόχο να αναπτύξουμε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Κυρία Επίτροπε, θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει το συντομότερο δυνατόν μια στρατηγική για τον Ατλαντικό. Μια στρατηγική η οποία θα περιλαμβάνει τη στρατηγική του 2020 για την ενέργεια και τη βιοπικιλότητα, για να καταπολεμήσουμε την αλλαγή του, του κλίματος και να προάγουμε μια αστική ανάπτυξη και μια βιώσιμη ανάπτυξη. Να βοηθήσουμε τον τουρισμό, τις έρευνες, τις καινοτομίες, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις θαλάσσιες μεταφορές και την εκπαίδευση. Για να βελτιώσουμε την πρόσβαση στις περιοχές μας μέσω της ανάπτυξης νέων θαλασσίων οδών. Να αναπτύξουμε νέες υποδομές και τεχνολογίες καθώς και τεχνολογία πληροφορικής και τηλεπικοινωνίας και ε, οργάνωση σε δίκτυα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Ευρωπαϊκό Όμιλο για την εδαφική συνεργασία, διότι έχει κάνει πολύ σημαντικές εργασίες για την ανάγκη να αναπτύξουμε τις ε, πολιτικές για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλέματος και να έχουμε μια ανάπτυξη πραγματικά βιώσιμη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η στρατηγική αυτή είναι υψίστη σημασία για τι περιοχέ του Ατλαντικού, αλλά όχι μόνο για αυτέ τι περιοχέ, αλλά για το σύνολο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τόιρερ για δύο λεπτά. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η στρατηγική της Βαλτικής ήταν το ενεκτήριο ελάχιστος η στρατηγική για τον Δονάβη, το δεύτερο βήμα και τώρα έχουμε την περιοχή του Ατλαντικού. Η ομάδα ΑΛΤΕ εδώ στο Κοινοβούλιο υποστηρίζει αυτή την περιφερειακή προσέγγιση και συνεργαστήκαμε ε, στην προετοιμαστία, βελτίωση των θαλασσών και προστασία του περιβάλλοντος, αλληλεία, θαλάσσια θάματα, αλλά περισσότερο τρεις πυλώνες στην εργασία των κρατών μελών για να εκμεταλλευτούν καλύτερες συνεργίες κατόπιν δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο ελληνικός συνδέει τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Ατλαντικό με άλλες χώρες υπερατλαντικά αλλά και με το, την Ισλανδία, το, την Ορβηγία, οπωσδήποτε βέβαια είπα και Καναδά. Και θα πρέπει να συνεργαστούν επίσης μεταξύ τους αυτές οι διάφορες περιφέρειες. Θα πρέπει να φροντίσουμε οι πόλεις, οι τοπικές αυτοδιοίτησεις, οι χώρες και οι πολίτες, η κοινωνία των πολιτών και οι επιχειρήσεις να δικτυωθούν ούτως ώστε όλοι οι παράγοντες ε, να μπορούν να δώσουν πνεύμα ζωή στην ε, αυτή πολιτική. Δεν πρόκειται δημιουργία νέων θεσμικών οργάνων. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα χρήματα που υπάρχουν. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχουν ίσως ακόμα ανοιχτέ δυνατότητες συνεργασίες ε, για την αντιμετώπιση των κοινών προβλημάτων και ακριβώς η ομάδα της Άλτε εδώ θεωρεί ότι υπάρχει δυνατότητα δράσης γιατί απειλείται το διεθνές εμπόριο γιατί πολλά από τα αγαθά της Ευρωπαϊκής Ένωσης έρχονται από τον Ατλαντικό και θα πρέπει να υπάρχουν και πολλές δυνατότητες εκμετάλλευσης των πρώτων υλών ίσως στον Ατλαντικό θα πρέπει όμως να προστατεύσουμε βιώσιμα την περιφέρεια αυτή και θα είναι, χαιρόμαστε που θα υπάρχει μια συνολική στρατηγική. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία Λεύεν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολλά χρόνια δεν είχαμε διαχειριστεί τις θάλασσές μας σωστά. Υπάρχουν διάφορα ε, συμφέροντα. ενέργεια, τουρισμός, αλληλεία, μεταφορές. Όλες οι στρατηγικές όπως για τον Ατλαντικό, το Δούναβι ή τη Βαλτική θα πρέπει να ορίσουν τους στόχους προτεραιότητας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ορισμένε πολιτικές αποφασίζονται σε κοινοτικό επίπεδο αλλά οι περιβαλλοντικές ε, ε, πολιτικές είναι θέμα των κρατών όλων με και γι' αυτό είναι καλό να υπάρχει μια ολοκληρωμένη ε, προσέγγιση για τον Ατλαντικό. Θα πρέπει να δώσουμε περιοριότητες στους διάφορους στόχους. Η συνεργασία με άλλες χώρες στην περιοχή του είναι επίσης πάρα πολύ σημαντική παραδείγματος χάρη θα πρέπει να μειωθούν τα πλαστικά απόβλητα, να καταπολεμηθεί η παράνομη ελεία και να ελέγχονται πολύ σωστά οι υπόλοιποι ελεείς. Όλοι εξαρτώμεθα με την υγεία μας από καλό και υγιές περιβάλλον. Όχι μόνο η ελεία και ο τουρισμός. Γι' αυτό οι περιβαλλοντικές στόχοι δεν αφορούν μόνο το περιβάλλον αλλά και την ευμάρεια στην περιοχή αυτή. Ευχαριστώ κύριο Βλάσακ, δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, όπως βλέπουμε, η στρατηγική, της, η της Βαλτικής αποτελεί πηγή έμπνευση κατά κάποιο τρόπο για άλλες περιοχές. Μετά τη στρατηγική του Δούναβη φτάνουμε σε μια στρατηγική για την περιοχή του Ατλαντικού. Μια πολύ συγκεκριμένη περιοχή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση για μεγάλο διάστημα αντιμετώπισε τον Ατλαντικό ως τα πλαίσια μιας διαμεθοριακής συνεργασίας. Η περιοχή του Ατλαντικού έχει στηριχθεί από το Interreg 3 β και εντάσσεται στην, στο υφιστάμενο πρόγραμμα ε, εδαφικής συνεργασίας στο πλαίσιο του στόχου 3. Στόχος εδώ είναι η προώθηση στρατηγικών ε, περιφερειακής ανάπτυξης σε διαμεθοριακό επίπεδο και να βελτιωθεί η πρόσβαση στην ε, κοινωνία της πληροφορίας, να προστατευθούν το περιβάλλον και οι φυσικοί πόροι και να ενισχυθούν οι οικονομίες των περιφερειών. Θα ήταν λοιπόν καλό να αξιολογηθούν τα υφιστάμενα προγράμματα και τα ωφέλη τους και μόνο τότε να αναπτυχθεί μια νέα στρατηγική για την περιοχή. Βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρέπει να συμπεριληφθούν και οι διατλαντικοί δεσμοί σε αυτή τη στρατηγική. Γιατί είτε μας αρέσει είτε δεν μας, αρέσει, είμαστε κομμάτι του ευρωατλαντικού χώρου και υπάρχουν αξίες στον ωκεανό αυτό. Ακριβώς όπως και η άλλη πλευρά της θάλασσας θέλουμε ελεύθερη διακίνηση των ε, προϊόντων του κεφαλαίου και των ανθρώπων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν αλληλοσυμπληρούμενες πολιτικές που συχνά δεν είναι συντονισμένες. Θα πρέπει να θέσουμε τις βάσεις για μια διατλαντική συνεργασία ως κομμάτι των πολιτικών τη Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό να συντονιστούν καλύτερα αυτά τα οποία κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην περιοχή του Ατλαντικού. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα φιλόδοξο πρόγραμμα που να μην περιορίζεται στα εθελοντικά μέτρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η κυρία Σβένσον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όταν μιλάμε για την περιοχή του Ατλαντικού, αναφερόμαστε σε δύο σημαντικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να επισημάνω αυτή τη στιγμή. Καταρχάς τα οικολογικά θέματα. Η βιωσιμότητα της αλληλείας είναι πολύ σημαντική και επίσης να δούμε τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν ε, δεν τηρούνται οι αλληλευτικές συμφωνίες, όπως γίνεται με την περίπτωση του Μαρόκου. Στην αλληλεία το 30% των ε, ζωνών επιτροπόμενης αλίευσης είναι κλειστά και ενώ φαίνεται να είμαστε μια περιοχή η οποία είναι πλούσια σε αλλιεύματα, εισάγουμε άνω του 30% των αλλιευμάτων. Και αυτό φυσικά έχει επιπτώσεις και σε φτωχότερες χώρες, διότι δεν έχουν πρόσβαση στις πρωτεΐνες που περιλαμβάνουν τα ψάρια και που βρίσκονται ε, σε αυτές τις περιοχές. Επίσης, τι γίνεται όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ανανεώνει, για παράδειγμα, συμφωνία, όπως ε, Για παράδειγμα συνέβη το 1975 όπου το Μαρόκο ε, εισέβαλε στην ε, Δυτική Σαχάρα και παρά το γεγονός ότι όλοι δήλωσαν ότι η περιοχή είναι υποκατοχή υπάρχουν επιπτώσεις για την αλία και τι γίνεται με τους κατοίκους της περιοχής. Όταν λοιπόν συζητάμε συμφωνίες θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και στοιχεία τέτοια αλλά πρέπει να λάβουμε και υπόψη στοιχεία βιωσιμότητας. Όπως σας λέω η στρατηγική αυτή είναι πολύ σημαντική και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να σέβεται τα δικαιώματα των λαών. Δεν μπορούμε να διατηρούμε, ε, για παράδειγμα, συμφωνία με το Μαρόκο, λαμβάνοντα υπόψη ότι υπάρχουν και συγκεκριμένε ε, εδαφικά προβλήματα στην περιοχή. Ο κύριο Κλάρκ. Εδώ γίνεται αναφορά σε άλλες πολιτικές όπως η κοινή ελληνική πολιτική και αυτό είναι φοβερό. Ποτέ δεν θα πρέπει να είχαμε σκεφτεί τέτοια πράγματα. Οι, οι Βρετανοί ε, ψαράδες έχουν περι, προστατεύσει πολύ προσεκτικά τα, τα αποθέματα αλλιευμάτων, αντιθέσει με τους άλλους. Βεβαίω πολλοί δεν, βλέπουν τη στιγμή να μπουν στη Βόρεια Θάλασσα. Θα πρέπει αποκλεισμό να υπάρχει, περισσότερο αποκλεισμό, όχι λιγότερο. πρέπει οι, ψαράδες φροντίζουν επί χρόνια, επί ε, ε, γενναίες ε, τα αποθέματα. Και εκεί υπάρχουν πλάσματα τα οποία αποτελούν τη βάση της τροφικής αλυσίδας. Αυτό αποτελεί την ζωή, το βιός των αλλιέων. Και τώρα πρόκειται να έρθουν, ε, να επιτραπούν μετακινήσεις ενός ε, ε, εκατομμυρίου τόνων χαλικιού στην περιοχή για τη δημιουργία μιας, ενός αιωλικού πάρκου στα νύχτα. Τι ζημιά θα προκαλέσει αυτό. Πόσο καιρό θα περάσει μέχρι ότου οι αλληλείς αναγκαστούν να κάθονται για να βλέπουν την καταστροφή των αλληλευμάτων τους. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μέλτσα. Ε, ο Ατλαντικός είναι πάρα πολύ σημαντικός και οικονομικά και οικολογικά για την Ευρώπη. Το ξέρουμε όλοι. Όσον αφορά την οικολογία ξέρουμε ότι ε, το ρεύμα του Μεξικού ε, έχει σημαντική επίδραση στο κλίμα της Ευρώπης. Το ποιε είναι οι αλλαγέ τα τελευταία χρόνια και τι θα γίνει στο μέλλον, βέβαια δεν ξέρουν καθόλου ούτε οι ίδιοι εμπεριγνώμοντες όσον αφορά την ε, ε, οικονομία θα πρέπει να δούμε κατά πόσον η Κολομβία και η Κίνα θα πραγματοποιήσουν την ε, συνδρομική σύνδεση Ατλαντικής και πλευράς και πλευράς του ελληνικού της Νοτιού Επίσης παίζει σημαντικό ρόλο για τα κύματα προσφύγων ο Ατλαντικός. Το 2005 παραδείγματο χάρη πολλοί άλλαξαν τις ζωέ και περνάνε μέσα των Καναρίων νήσων στον Ατλαντικό. Όλα αυτά έχουν σημαντικές επιπτώσεις. Τους επόμενους μήνες θα μπορούν ε, οι πρόσφυγες που έχουν φτάσει στις, δεκα, στις δεκάδες χιλιάδες ε, που υπάρχουν ήδη ε, ενώ οι πρόσφυγες στις ακτές της Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι ένα τίποτα σχετικά με αυτό που μας περιμένει. Θα πρέπει βέβαια να ισχύει η αρχή ότι οι πρόσφυγες θα πρέπει να τοποθετούνται κατά τον κοντά στις πατρίδες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζει ανακοίνωση για τη στρατηγική για τον Ατλαντικό, μια περιοχή που έχει δύο πολύ σημαντικές πτυχές και το γεγονός ότι είναι ένας ωκεανός και δεύτερον είναι ένας υπερπεριφερειακός τομέας. Μας ενδιαφέρει η διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ε, τα όσα σχετίζονται με τη θάλασσα και ο τουρισμός και γενικώ υπάρχουν πολιτικές οι οποίες είναι πολιτιματικές. Μας ενδιαφέρει επίσης το θέμα των μεταφορών, η λεγόμενη διασύνδεση και με τις περιοχές που βρίσκονται κατέρωθεν του Ατλαντικού, αλλά και με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση οι θαλάσσιοι αυτοκινητόδρομοι, ε, οι υπεροβολητικές συνθήκες. Αυτά όλα θα πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα. Στη Γαλλικία, ε, στην περιφέρειά μου, ε, υπάρχουν και περιοχές που μπορούν να συνδεθούν και με την Πορτογαλία. Και δεν θα πρέπει να επικεντρωθούμε μόνο σε θαλάσσια θέματα. Όπω έλεγε και ο κύριο Καντέκ, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την πολύ σημαντική εδαφική διάσταση διότι μπορούμε να έχουμε ε, εδαφική, οικονομική και κοινωνική συνοχή. Η στρατηγική θα πρέπει να σχετίζεται στενά με την στρατηγική για το 2020, την περιφερειακή πολιτική και τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές. Εν τέλει, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τους ε, διάφορους οργανισμούς και οργανώσεις που υπάρχουν ήδη για τον Ατλαντικό, Υπάρχει η οργάνωση της Γαλλικίας και η Ευρωπεριοχή που έχει ε, σχηματιστεί με την ε, Βόρεια Πορτογαλία που ήταν μία από τις πρώτες οργανώσεις ε, εδαφικής συνεργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει μόνιμο διάλογο και με τις οργανώσεις αυτές και τις περιφέρειες και για την εκπόνηση στρατηγικής αλλά και για τη μελλοντική της εκτέλεση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Γκρελία, για ένα λεπτό. Κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, χαίρομαι για αυτό το σχέδιο στρατηγικής για την περιοχή του Ατλαντικού. Έχουμε ανάγκη μια τέτοια προσέγγιση για τη θαλάσσια περιοχή λόγω της ιδιαιτερότητας και βεβαίως ε, των προβλημάτων της. Συγκεκριμένα ως εκλεγμένη της Νορμανδίας θέλω να επιστήσω την προσοχή σα ε, στην ιδιαιτερότητα της μάχης και στα πλαίσια της στρατηγικής του Ατλαντικού. Η στρατηγική προσέγγι, θαλάσσια προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Ατλαντικό και τη Βόρεια Θάλασσα ε, πρέπει να λάβει υπόψη ότι ένα μεγάλο ποσοστό των πλοίων ε, περνούν από την περιοχή. Εκεί υπάρχει αλληλεία, ψυχαγωγία και πολύ σύντομα θα υπάρχει και ε, προς μεγάλη μου χαρά παραγωγή ενέργειας χάρη στην, στα θαλάσσια ολικά πάρκα. Πρέπει λοιπόν να ληφθούν όλα αυτά υπόψη τους να αναλυφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όλα αυτά να γίνουν στα πλαίσια μιας στρατηγικής του Ατλαντικού και βεβαίως η... Ε, ε, σας έχω αναφερθεί, έχω αναφερθεί κυρία ε, Επίτροπε στο θέμα αυτό της κοινή χρηματοδότησης και στο παρελθόν σε εσάς κυρία Επίτροπε. Κοιτάξτε, υποστηρίζω ό,τι γίνεται στην ευρωπαϊκό επίπεδο για την ε, ο, συντονισμένη προσέγγιση. Πέντε χώρες ε, του, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ακτές στον Ατλαντικό. Δηλαδή το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Πορτογαλία και η Ισπανία. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να συμπεριληφθούν και η Νορβηγία, η Ισλανδία και η Νήσι Φερόες οποιαδήποτε στρατηγική θα πρέπει η στρατηγική να εστιαστεί στην ε, οικονομική ανάπτυξη. Ε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν και περιοχές που δεν έχουν ανεπτυγμένη παραγωγή ενέργειας, παραδείγματο χάρη. Το 50% θα μπορούσε να, στο μέλλον να τροφοδοτείται η ε, ανάγκες ε, ενέργειας Ευρωπαϊκής Ένωσης από ανανεώσιμες πηγές ε, στις ε, πλές του Ατλαντικού. Υπάρχει ένα τεράστιο δυναμικό ανάπτυξη στην περιοχή αυτή, σε συμπληρωμένη στις αναπτυκτής στρατηγικά τοποθετημένων ε, λιμένων μαρίνας, δηλαδή στην περιοχή αυτή. Επίσης όσον αφορά την ηχθειοκαλλιέργεια, την υδατοκαλλιέργεια, στενή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, καθ' όλο το μήκος του Ατλαντικού. Η στρατηγική του Ατλαντικού θα πρέπει να ε, εξεταστεί βέβαια και μέσα στα πλαίσια της κοινή αλληλευτικής πολιτικής γιατί στο Ανατολικό υπάρχουν τα πιο πλούσια αλληλευτικά υδατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης υπάρχουν εκεί οι τόποι στους οποίους παράγονται πάρα πολλά είδη θα πρέπει να είναι βελτιωμένη η εποπτεία και η προστασία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μία ε, ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εξασφαλίσει καλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Και αυτό κύριε Πρόεδρε θα οδηγήσει σε καλύτερη απάντηση σε περίπτωση ε, υποθέσεων πρώτης ανάγκης και επίση θα δοθεί η δυνατότητα καταπλέμησης οργανωμένου εγκλήματο και λαθρεμπορίου εναρκωτικών. Ευχαριστώ ε, κύριε Τσανέσκι. Κυρίε και κύριοι, η προφορική ερώτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στρατηγική για την περιοχή του Ατλαντικού είναι ένα περαιτέρω βήμα και καταδεικνύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναπνέει από διαφορετικούς πνεύμονες. Έχουμε τη στρατηγική για το Δούναβι, η οποία είναι πρωτοβουλία της ε, Ουγγρικής Προεδρίας και τώρα η η ώρα για την ε, περιοχή του Ατλαντικού η οποία άπτεται πέντε ευρωπαϊκών χωρών αλλά είναι πάρα πολύ σημαντική διότι δεν μπορεί να αποτελέσει απλώς ε, τρόπο για να αυξηθούν οι πόροι της χώρας ε, των χωρών που ε, βρίσκονται στον, Ατλαντικό, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται και καλύτερα οι περιοχές αυτές. Η κυρία Ρόσμπαχ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εάν η προστασία του θαλάσσιου περι, ε, περιβάλλοντος είναι ε, βασική στρατηγική στο θέμα αυτό ή θα σταθείτε ε, στο θέμα των απορριμμάτων πλαστικών στις θάλασσες και στην περιοχή του Ατλαντικού πιο συγκεκριμένα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εξετάσει το θέμα της ε, παράνομης αλληλείας και την ε, εσκεμμένη απόρριψη ε, πετρελαίου. Μπορούν να ληφθούν υπόψη αυτά τα στοιχεία στη στρατηγική. Υπάρχουν και το θέμα των κρουαζιερόπλων και η ρήπανση των θαλασσών που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Η Επίτροπος θα ασχοληθεί και με τις θαλάσσιες οδό, οδούς που συμπεριλαμβάνονται στη στρατηγική αυτή. Αν θέλουμε να μειώσουμε τη ρήπανση και τα απορρίμματα τα οποία μολύνουν τις θάλασσές μας, είναι πολύ σημαντικό να τα λάβουμε και αυτά υπόψη. Ο κύριος Τεξέιρα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Η συνθήκη της Λισαβόνας περιλαμβάνει τη ε, εδαφική συνοχή και αυτό είναι πολύ σημαντικό και για την περιφερειακή μας πολιτική. Για να είναι αποτελεσματικές οι πολιτικές μας θα πρέπει να έχουμε και νέες στρατηγικές για τις περιοχές της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και για να είναι επιτυχής οι στρατηγικές αυτές θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιοχή που θα βασίζονται στις ιδιωτερότητες και τα συγκεκριμένα προβλήματα που βιώνει κάθε περιοχή. Η περιοχή του Ατλαντικού έχει πολύ συγκεκριμένε ιδιαιτερότητε που πρέπει να περιληφθούν σε μια φιλόδοξη πολιτική. Υπάρχουν περιοχέ οι οποίε είναι απομακρυσμένε και έχουν προβλήματα σύνδεση. Επίση είναι πάρα πολύ ευάλωτη περιοχή και αποδυναμώνεται συνεχώ από τι αλλαγέ του κλίματο. Επίση, υπάρχουν ε, πολύ εντατικές ε, θαλάσσιες δραστηριότητε και λόγω μεταφορών αλλά και λόγω δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την αλληλεία και την ενέργεια. Στην περιοχή του Ατλαντικού περιλαμβάνονται και υπερπεριφερειακές ε, ε, περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, η ολοκληρωμένη λοιπόν στρατηγική για τον Ατλαντικό θα πρέπει να λάβει υπόψη της όχι μόνο τη μεγάλη θαλάσσια στρατηγική αλλά και μια μεγάλη εδαφική ε, συνιστόσα. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε η στρατηγική αυτή να έχει και επιπρόσθετο έθελος ε, για την ε, περιοχή, να λάβουμε υπόψη όλες τις περιοχές, αλλά και τις υπερπεριφερειακές περιοχές της Μαδέιρας, των Αζωρών και των λοιπών περιοχών, και να λάβουμε υπόψη ότι λόγω των ε, γεωγραφικών ε, και διαρθρωτικών διαφορών που έχουν θα πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια πολιτιομερική διακυβέρνηση στη στρατηγική αυτή και οι τοπικές και περιφερειακές αρχές θα πρέπει να συμμετέχουν ήδη από το σημείο της διάγνωσης της περιφερειακής πραγματικότητας μέχρι την εκπόνηση της στρατηγικής. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θέλω πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον κύριο Καντέκ για την εξαιρετική αυτή πρωτοβουλία του που σκοπό έχει την εκπόνηση μιας στρατηγικής του Ατλαντικού που σαφώς τη χρειαζόμαστε στο μέλλον. Αυτό είναι σαφές και από όσα είπαν οι προλαλήσαντες. Μιλάμε για μια συγκεκριμένη, ιδιαίτερη περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αλληλεία, οι μεταφορές, αλλά και όλα τα άλλα θέματα πρέπει να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά και αυτό μπορεί να γίνει στο πλαίσιο μιας γενικής στρατηγικής για τον Ατλαντικό. Η περιφερειακή συνεργασία είναι κάτι που στηρίζεται από το 1990. Ένα μέρος του Ταμείου Συνοχής έχει χρησιμοποιηθεί για αυτό το σκοπό. Οι διάφορες αυτές στρατηγικές γεννήθηκαν στα πλαίσια της Σουηδικής Προεδρίας. Ελπίζω ότι θα αυξήσουν τη διαμεθοριακή συνεργασία και στο μέλλον η συνεργασία στον τομέα της ενέργειας, των μεταφορών και των επιχειρήσεων οπωσδήποτε μπορούν να αναπτυχθούν στα πλαίσια τέτοιων στρατηγικών. Όπως επισημαίνει η πρόταση το σχέδιο ψηφίσματος, η στρατηγική αυτή, όπως και οι άλλες, θα πρέπει να στηριχθεί στις υφιστάμενες στρατηγικές και στην υφιστάμενη χρηματοδότηση. Δεν χρειάζεται να αναπτυχθούν νέες δομές για την περιοχή του Ατλαντικού όλες οι περιφέρειες και όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για να απτυχθεί η δυνατή, καλύτερη δυνατή συνέργεια. Ευχαριστώ, ο κύριος Κέλλη. Σας ευχαριστώ που δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσω για το σημαντικό αυτό θέμα. We have seen the Danube, the Baltic, the Mediterranean strategies είναι σημαντικό ο συνδυασμός των στρατηγικών ε, γιατί όπως είπανε πολλοί υπάρχει τεράστιο δυναμικό και ιδίω υπάρχει ο θαλάσσιος τομέας αλλά και ο δαφικός τομέας όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως. Εγώ θα ήθελα να τονίσω δύο πτυχές τουρισμό και ενέργεια. 7% του Ιρλανδικού τουρισμού βασίζεται στον Ατλαντικό. Και θα πρέπει να προσπαθήσουμε μέχρι το 2020 να διπλασιάσουμε αυτό το ποσοστό. Σε όλες τις πέντε χώρες που έχουν ε, ακτές στον Ατλαντικό. Υπάρχουν πολλές δραστηριότητες τουριστικές ε, περίπατος, υποβρύχια αλία, αλία γενικά, σερφ. Θα πρέπει να υπάρχει ενοποιημένη προσέγγιση όλων των εκεί περιοχών. Μειώντα και την γραφειοκρατία θα έλεγα. Όσον αφορά τώρα την ενέργεια, το 2050 θα χρειαζόμαστε πολύ περισσότερες ε, ε, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από ό,τι σήμερα ο Ατλαντικός ωκεανός με την ε, παλήρια, με τον άνεμο έχει πολύ μεγάλο δυναμικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Uh, ο Άλβες, ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναπτύξει μία στρατηγική για τον Ατλαντικό για να αναπτύξει τις δυνατότητες που έχει αυτή η τόσο προνομίουχα περιοχή που μας ενώνει με πολύ σημαντικές περιοχές του κόσμου όπως η Βόρεια Αμερική, η Νότια Αμερική αλλά και σημαντικές πλευρές της Αφρικής. Μόνο μέσω μιας στρατηγικής για, για τον Ατλαντικό μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις δυνατότητες και να υπάρχει προστιθέμενη αξία όχι μόνο για τις περιοχές αυτές αλλά και για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με έναν ενωμένο στρατηγικό προσανατολισμό μπορούμε να κάνουμε αυτές τις παράκτης περιοχές λιγότερο περιφερειακές, πιο κεντρικές και ε, συγχρονισμένες με τους υπολείπους μια στρατηγική για τον Ατλαντικό στην οποία θα συμμετέχουν όλα τα κράτη-μέλη της περιοχής ε, και από εδαφικής πλευράς θα μας επιτρέψει να έχουμε ανάπτυξη και σε οικονομικό και σε επιστημονικό τομέα ε, και να προσέξουμε ιδιαίτερα θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον, με τις επιστημονικές ε, εξελίξεις, με προϊόντα τεχνολογίας, τα ΕΦΗ προηγόντα. Η κυρία Ερικογέν Πέρες, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, βιώνουμε μια πολύ σημαντική ε, στιγμή για την ε, ε, πολιτική συνοχή, η οποία από την έναρξη ισχύα τη συνθήκη τη Λισαβόνα δεν επικεντρώνεται μόνο στι οικονομικέ και κοινωνικέ πτυχέ, αλλά έχει και μια εδαφική συνιστόχα. Η εδαφική συνοχή προποθέτει αρμονική συνύπαρξη μεταξύ των εδαφών, ώστε οι πολίτε να μπορούν να εκμεταλλευτούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τι εδαφικέ ιδιαιτερότητέ του. Επίσης, είναι απαραίτητο να υπάρξει πρόεδρος ε, στη συνεργασία μεταξύ των περιοχών της Ένωσης που αντιμετωπίζουν τις ίδιες προκλήσεις και, τους ίδιους προβληματισμούς. Αυτό είναι ο στόχο ε, τη Στρατηγική Ευρωπαϊκή Ένωση για την περιοχή του Ατλαντικού. Μια κοινή προοπτική για να αντιμετωπίσουμε τι κοινέ προκλήσει που αντιμετωπίζουν οι χώρε τη περιοχή. Μεταξύ άλλων, οι θαλάσσιες έρευνες, ε, η παρακολούθηση των θαλασσών και οι οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις. Για να επιτύχουμε τους στόχους μας θα πρέπει να υπάρχει στρατηγική, ολοκληρωμένη ε, πολιτική η οποία θα συνδυάζεται με την στρατηγική του 2020 και τις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις δημοσιονομικές προοπτικές για μετά το 2013 και να λάβουμε υπόψη και τη θαλάσσια πολιτική. Κυρίες και κύριοι όμως, πρωτίστως θα πρέπει η στρατηγική αυτή να έχει μία πολυεπίπεδη διακυβέρνηση η οποία θα βασίζεται στη με πιο στενή συμμετοχή των τοπικών, ε, περιφερειακών και εθνικών αρχών και τους ενδιαφερομένους από τον ιδιωτικό τομέα, καθώς επίσης και τις οργανώσεις Κοινωνία κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων και των ε, διεθνών ε, οργανώσεων που συμμετέχουν στα αντίστοιχα δίκτυα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η διαδικασία κατστιάει τώρα. Η κυρία Πατράο Νέβες, καταρχάς, για ένα λεπτό. Ε, ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Ένας είναι ο στόχος της ε, στρατηγικής αυτής. Να αντιμετωπίσει τους ωκεανούς και τις θάλασσες της Ευρώπης με ενοποιημένο τρόπο αλλά και ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές τους. Υπάρχει μεγάλη πολυμορφία και η περιοχή αυτή είναι μια απομακρυσμένη και βαθύτερη περιοχή. Έχει και ιστορικές ε, ρίζες και με τις δύο πλευρές του Ατλαντικού και γι' αυτό πρέπει πραγματικά να αντιμετωπιστεί χωριστά. Είναι μια γεωστρατηγική περιοχή μεταξύ Ευρώπης, Αμερικής, Αφρικής και υπάρχουν διάφορες δραστηριότητες. Πρέπει επίσης να προστατευτούν τα οικοσυστήματα, να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή και να υπάρχει προμήθεια τροφίμων και ενέργειας. Είναι μια περιοχή πλούσια σε πολλών ειδών πόρους. Δεν θεωρούμε λοιπόν ότι πρέπει να υπάρξουν θα πρέπει να υπάρξουν λοιπόν προγράμματα έρευνας και τεχνολογίας για την βιώσιμη χρήση αυτών των ε, πόρων. Χρειάζεται λοιπόν στις Αζόρες θα έλεγα εγώ ένα παρατηρητήριο ε, ανοιχτής θάλασσας. Ευχαριστώ. κύριε Σμίθ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι συμφωνεί η Κομισιόν και, ε, το, και εμείς ε, για τη στρατηγική αυτή και πιστεύω ότι θα, θα πετύχουν πολύ περισσότερα με τη δημιουργία ενός φόρουμ το Συμβούλιο θέτει προτεραιότητες και αυτό μας πλήττει. Αν θέλουμε λοιπόν να πετύχουμε 300 εκατομμύρια στόχους, ίσως να μην πετύχουμε τίποτε. Θέλω λοιπόν να θέσω ε, δύο προτεραιότητες όπου μπορεί να προσθεθεί αξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτον, η, αγωγή σύνδεσης για την θαλάσσια ενέργεια υπάρχει τεράστια ποσότητα στη Σκωτία και μπορεί αυτό να παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Η παράγραφη 9 11 η σημασία της των θαλασσίων μεταφορών μπορεί να έχει τεράστιο όφελος και για την οικονομία και για το περιβάλλον. Πολλά πρέπει να θαυμάσουμε εδώ, αλλά ελπίζω ότι η Κομισιόν θα είναι πιο στοχευμένη ε, στους στόχους της. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ευχαριστώ. Θέλω να εκφράσω την πλήρη υποστήριξή μου στην ανάπτυξη όλων των θαλασσιών περιοχών. Οι ωκεανοί αποτελούν ευκαιρία για την ανάπτυξη των μεταφορών, της αλίας, της ενέργειας και της έρευνας οι ευκαιρίες διαχείρισης που ανοίγονται πρέπει να χρησιμοποιηθούν με φρόνηση, δεδομένου ότι η κοινότητα μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο του φύλακα, θεματοφύλακα του περιβάλλοντος. Ο Ατλαντικός ωκεανός είναι μια φυσιολογική διέξοδος οικονομικής ανάπτυξης. Οι θαλάσσιες μεταφορές αποτελούν, απαιτούν από εμά να δημιουργηθεί μια καλύτερη στρατηγική για την περιοχή αυτή και για τις λιμενικές εγκαταστάσεις, γιατί η θάλασσα ανοίγει τις πύλες στην Ενωμένη ΕΕ. Ευρώπη. Η κυρία Σάντσο Σμίθ έχει το λόγο. Merci, Monsieur le Président. Madame la Commissaire, chers collègues. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Από το 2005 το θέμα της περιφερειακής ανάπτυξης που ξεκίνησε από τη περιοχή της Βαλτικής συγκεντρώνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο Κοινοβούλιο. Χαίρομαι που σήμερα χάρη στον συνάδελφο Αλέν Καντέκ μπορούμε να έχουμε φιλοδοξίες για μια περιφερειακή πολιτική για τον Ατλαντικό. Πέρα από το συντονισμό και τις συνέργειες και τις σημασίες μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για να αντιμετωπιστούν τα χωροταξικά θέματα. Θέλω να επισημιστήσω την προσοχή σε δύο θέματα. Η εδαφική ε, συνεργασία, το σημείο 3 της πολιτικής συνοχής πρέπει να στηρίξει αυτή τη στρατηγική με τον συντονισμό των σκέψεων, των καθορισμών και το εύρος των προγραμμάτων. Θα πρέπει μέσα από τα επιχειρησιακά προγράμματα τα κράτη της περιοχής να συμμετάσχουν σε ε, κοινέ ε, ενέργειες. Χωρίς αυτό οι στρατηγικές αυτές θα παραμείνουν νεκρογράμματα. Αν δεν θέλουμε να ε, δημιουργήσουμε μεγάλες περιοχές θα αποδείξουμε ότι δεν έχουν εξαφανιστεί τα σύνορα. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Δαμανάκη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έγινε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση και έχει αποδειχθεί ότι η πρωτοβουλία αυτή της ε, προφορικής ερώτησης ήταν επιτυχημένη. Τρία σημεία κύριε Πρόεδρε. Πρώτον, όσον αφορά τη θελάσσια στρατηγική μας σε αυτήν μπορούμε να συμπεριλάβουμε πολλούς τομείς, πολλές δραστηριότητες και να δοθούν πολλές προοπτικές. Πού θα επικεντρωθούμε. Θα επικεντρωθούμε στην προσπάθεια να δημιουργηθούν επαφέ επαφές ανάμεσα στους διάφορους τομείς. Δηλαδή, υπάρχει ένα χώρος, ένας θαλάσσιος χώρος, ο χώρος του Ατλαντικού. Εκεί μπορεί να υπάρξει αλληλεία, χρειάζεται προστασία του περιβάλλοντος, μπορεί να υπάρξει τουρισμός, μεταφορές, ε, υδατοκαλλιέργειες, ενέργεια, έρευνα. Χρειάζεται λοιπόν να βρούμε έναν τρόπο να δημιουργηθούν σχέσεις μεταξύ όλων αυτών των, τομέων και να ξεπεραστούν οι τυχόν, τα τυχόν συγκρόμενα συμφέροντα. Άρα ο σχεδιασμός θα αποτελέσει ένα πολύ βασικό εργαλείο. Επίσης η παρακολούθηση η επιτήρηση αυτής της θάλασσας αλλά και η γνώση για τη θάλασσα θα αποτελέσουν σημαντικά εργαλεία. Αυτή είναι η φιλοδοξία μας. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε νέους, νέες δομές. Συμφωνώ με αυτό. Δεν χρειάζονται νέες δομές. Αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι σχέσεις, επαφές ανάμεσα στις υφιστάμενες δομές. Και περί αυτού πρόκειται δημιουργία επαφών, σχέσεων ανάμεσα στις υφιστάμενες δομές για καλύτερα αποτελέσματα. Το πρώτο μου θέμα ήταν αυτό. Το δεύτερο αφορά αυτό το οποίο είπατε ε, σε σχέση με μια ε, πολιτική εδαφική συνοχής. Σας υπενθυμίζω ότι υπάρχει αυτή η πολιτική για να υπάρξει μια πολιτική μακροπεριφερειακή πρέπει να υπάρξει πρόταση από το Συμβούλιο προς την Κομισιόν. Προς το παρόν αυτό το οποίο έχουμε είναι μια πρόταση για μια θαλάσσια στρατηγική. Ελήφθη τον περασμένο Ιούνιο απόφαση γι' αυτό ήδη έχουμε την εξουσιοδότηση να προβάλλουμε μια θαλάσσια στρατηγική. Το κάνουμε και ελπίζουμε ότι με αυτόν τον τρόπο βοηθάμε για να τεθεί επιτάπητος η ε, προοπτική μιας μακροπεριφερειακής προσέγγισης. Τρίτο σημείο. Υπάρχει ανάγκη για μια διεθνή προσέγγιση. Συμφωνώ με όλους όσοι ανέφεραν ότι χρειάζεται καλός συντονισμός με τους γείτονες και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να γίνουν καλές συζητήσεις και να, και να καθορίσουμε ε, ίδιους κανόνες για όλους, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να πετύχουμε. Για μία ακόμα φορά λοιπόν θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Καντέρ και την πρωτοβουλία του και θέλω να σας ε, διαβεβαιώσω ότι όλες οι προτάσεις σας θα ληφθούν υπόψη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κυρία Επίτροπε. Έχουμε ένα, μία πρόταση ψηφίσματος για να κλείσει η συζήτηση, η οποία τώρα έληξε. Η ψηφοφορία θα γίνει την Πέμπτη της στις 11.30. Ευχαριστώ όλους και τώρα θα περάσουμε...